Ευχαριστώ, Ζαν. Καλημέρα σε όλους. Όπως έχουμε πει στην πρώτη ανταλλαγή απόψεών μας, συμφωνούμε με την ε, βασική αντίληψη για το InvestEU και παρόλο που είχαμε βελτιώσει τις επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε ακόμη καλύψει το κενό που υπάρχει στις επενδύσεις. Οπότε υπάρχουν πολιτικές ανάγκες εξυγχρονισμού της δομής της οικονομίας μας για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει κενό επενδύσεων που μας έχει μείνει σπακαταθήκη του παρελθόντος, αλλά υπάρχει και κενό στις επενδύσεις ως μια ανάγκη για το μέλλον της οικονομίας μας. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την ιδέα να υπάρξει ένας νέος κύκλος συγκεκριμένων εργαλείων υποστήριξης των επενδύσεων. Συμφωνούμε με τα βασικά στοιχεία της πρότασης, ιδίως την απλούστευση και ευθυγράμμιση τη στήριξη των επενδύσεων, με τη δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου, ενός ενιαίου πλαισίου, όπου θα συνδυαστούν τα υπάρχοντα προγράμματα αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων, αλλά θα διευκολυνθεί και η πρόσβαση των δικαιούχων. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα ποσότητας. Αυτό θα τα αφήσω στον φίλο μου, τον Ζωζέ Μανουέλ. Υπ' αυτήν την άποψη συμφωνούμε ότι είναι καλή ιδέα το InvestEU να μπορέσει να διατεθεί και σε άλλους συνεργάτες εκτός από την Τράπεζα Επενδύσεων και το είπαμε και στις διαπραγματεύσεις μας για την πρόταση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει ένας αφέστερος ορισμός του 75% που θα διατίθεται στον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Εγγύηση και επίσης να αποσαφινιστούν οι συνεισφορές του ε, τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλων ε, οδοτήτων ως μέρος των δυνατοτήτων. Πρέπει να δούμε βέβαια τι θα ορίσουμε ως implementing partners, ποιοι θα είναι αυτοί οι συνεργάτες, εταίροι που θα εφαρμόζουν ε, για να μην υπάρχει μόνο ένας μεγάλος και υπάρχει βελτίωση σε αυτή την προσέγγιση αλλά δεν προβλέπονται ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν αλλάζουν τα βασικά στοιχεία και συστατικά. Λίγο πιο ριζοσπαστικοί θα είμαστε στην ομάδα προγραμματισμού που επιλέγει τα έργα. Καλύτερα είναι να μην υπάρχει αυτό το σώμα και αυτοί οι συνεργάτες που θα αναλαμβάνουν την υλοποίηση να αποτιμούν, να αξιολογούν το έργο. Όμως θα υπάρχει μια κοινή ε, μεθοδολογία και ένα scoreboard, ε, ένα βαθμολόγιο που με καταξιοδότηση πράξη θα το κοιτάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με τις τροπολογίες μας θέλουμε να βελτιώσουμε και τη λογοδοσία ε, έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το Διοικητικό Συμβούλιο, το Steering Board με προσώπους των κρατών μελών, του Κοινοβουλίου, των ε, συνεργατών, ε, θα καταρτίζονται κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχει βεβαίως διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το Steering Board. Υπάρχει και το, το Συμβούλιο ε, που έχει συμβουλευτικό ρόλο, όπου και τα δύο όργανα θα μπορούν να συνδυαστούν σε, μια κοινή, σε ένα κοινό σχηματισμό υπάρχει διάκριση μεταξύ των διαφορών ε, σχημάτων συνεδρίασης και επίσης θα μπορούσαν και επιτόπου εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στην επιλογή των έργων και προγραμμάτων για να μην υπάρχουν αντιφάσεις. ή παρατυπίες καθώς τα συνδυάζονται μεταξύ τους τα διάφορα προγράμματα και έργα. Σε ό,τι αφορά το σκέλος των 100 μελών, Ξέρετε ότι υπήρξαν ε, αμφιλεγόμενε απόψεις εδώ. Ε, θεωρούμε θετική τη δυνατότητα, που είναι απλώ δυνατότητα, πρόσθετη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη, να ε, ασχολούνται με το συνδυασμό, το blending των προγραμμάτων για να συνδυάζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο και στο υπάρχον σκέλος των Ταμείων Συνοχής. Και προβλέπουμε και τη δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν με τις ίδιες διατάξεις που προβλέπουν την ε, κατά περίπτωση εξέταση των ε, προσφορών αυτών με την πλατφόρμα του ΕΦΣΥ. Θα υπάρχει και η αξιολόγηση κινδύνου των ε, διάφορων δράσεων που θα προβλέπονται μέσα από τις προτάσεις των κρατών μελών και θα πρέπει να ορίζονται και οι όροι τη παραχώρηση και τα κίνητρα, ιδίω εκεί όπου είναι πιεστικέ οι συνθήκε τη αγορά. Πρέπει να προβλέπονται βιώσιμα προγράμματα και έργα, προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένε ελλείψει και κενά. Από ό,τι έχει δείξει η εμπειρία μας από τα διάφορα συμμετρικά σοκ. Επίση, θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή ότι σε όλε τι περιπτώσει με τι τροπολογίε μα θέλουμε να δίνουμε προσοχή στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στην ε, έκθεση έχουμε προβλέψει όλα αυτά τα στοιχεία και τα έχουμε συνδυάσει με τα κριτήρια επιλεξιμότητα ε, για να εντοπίζονται και οι συνεργάτες που θα υλοποιούν. Ε, είμαστε στη διάθεσή σας λοιπόν για τις παρατηρήσεις σας για να δούμε με τροπολογίες θα τις καλύψουμε. Ευχαριστώ Ρομπέρτο, ο Ζωζε Μανουέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ξέρουμε, το InvestEU έρχεται να αντικαταστήσει όλα τα δημοσιονομικά εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τα χρηματοδοτικά λοιπόν μέσα και εδώ πρέπει να δούμε πως το ερχόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα μειωθεί το επίπεδο σε σχέση με το σημερινό. Δεν έχει καμία λογική η εγγύηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρηματοδοτικά εργαλεία να μειωθεί από το 2021 στο 2027. Και αν δούμε τι γίνεται με το, ταμείο, ε, το κονδύλι για την εγγύηση που προκλείται αυτή τη στιγμή για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και κοιτάξουμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτό το χρηματοδοτικό μηχανισμό του InvestEU από το 2021 στο 2027, βλέπουμε ότι υπήρξε μείωση Γι' αυτό λοιπόν όχι στην έκθεση αυτή, αλλά στην έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα κοιτάξουμε με μια τροπολογία να προσπαθήσουμε να παρέμβουμε για να ενισχύσουμε το Ταμείο τη Εγγύηση για, με 1.200 εκατομμύρια ευρώ για να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο το 2021 με 27, συγκρίνοντας με το 2014-2020. Η κατάσταση αυτή, μάλλον η πρόταση αυτή, νομίζω ότι την τη συμφωνία όλων και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αλλάξει το επίπεδο εγγύηση για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα που καταστήσουν όλα τα προηγούμενα. Είναι προφανέ ότι αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, το InvestEU, θα πρέπει να συμφωνεί με τις πολιτικές, τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συμφωνίες που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές τις οποίες έχει αναλάβει δεσμεύσεις, όπως τη Συμφωνία των Παρισίων, και όλους τους στόχους ε, και σκοπούς που έχουμε αναλάβει, όπως τους στόχους της χιλιετίας. Όλε οι συμφωνίε λοιπόν, τι οποίε έχουμε συνάψει, θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ. Προκειμένου να εγκριθούν τα έργα και τα προγράμματα μέσω του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου. Το InvestEU δεν έρχεται να αποκαταστήσει ούτε θα αντικαταστήσει την πολιτική συνοχή. Πρέπει όμω να συνεισφέρει για την οικονομική συνοχή, για την κοινωνική συνοχή, για την εδαφική συνοχή. Ε, υπάρχουν τροπολογίε που ε, επιδιώκουν αυτόν τον στόχο. Θέλουμε να υπάρχει εδαφική ισορροπία και μέσα από τις επενδύσεις. Η πρόταση αυτή λοιπόν θέλει να ενισχύσει τις περιοχές που υπάρχουν καθυστερήσεις, να υπάρχουν έργα εκεί, σε περιοχές με ε, δυσκολίες, με δυσχέρειες. Για κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, δημοσιονομικούς φορείς, ε, χρηματοδοτικούς φορείς μάλλον, για να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για νεοφυείς εταιρείε, για τα διπλώματα και, και την καινοτομία. Αυτό με τις τροπολογίες μας. Εδώ λοιπόν το συμβούλιο που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, το advisory board, δεν έχει κανένα νόημα να αποτελείται μόνο από μέλη των κρατών μελών και να υπάρχει άλλο από τα χρηματοπιστωτικά ή τι αναπτυξιακέ τράπεζε ή τι τράπεζε επενδύσεων. Θα πρέπει όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε διάλογο. Δεν θέλουμε να τους βάλουμε ξεχωριστά του εκπροσώπου των κρατών μελών, των αναπτυξιών τραπεζών και όσων θα συνεισφέρουν, αυτού που θα αναλάβουν τα έργα. Ενισχύουμε το ρόλο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που θα μπορεί για, την κάθε μια, για, το καθένα από τα τέσσερι, για την κάθε μια από τις τέσσερις θηρίδες, τις τέσσερις κατηγορίες, να ορίσει δικαιούχους που θα μπορούν να υποφεληθούν και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν. Και υπάρχει και μια διεύρυνση ως προς το ποιοι θα είναι επιλέξιμοι ως ε, δικαιούχοι. Ενισχύεται και ο ρόλος του Κοινοβουλίου με το Steering Board και επίσης με λογοδοσία, με το πώς ελέγχονται τα κονδύλια. Γιατί θα υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις, investment guidelines, κάτι που θα αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προασπίζομαι το σκέλος του 5% για τα κράτη-μέλη. Είναι ε, θελούσια η συνεισφορά. Βέβαια υπάρχει μεγάλη διστακτικότητα και από την Επιτροπή της Περιφερειακής Ανάπτυξης και από αρκετούς συναδέλφους. Όμως αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με όσα γίνονται και έχει επικριθεί, έχει τύχει πολλών επικρίσεων την ε, μεταφορά του Ταμείου Συνοχής για το για τη διευκόλυνση διασύνδεση της Ευρώπης στο ΣΕΦ. Εδώ υπάρχει δυνατότητα σε ένα μέγιστο όριο 5% τα κράτη-μέλη να πάρουν το 5% των διευθυντικών ταμείων και να το πάνε σε αυτό το σκέλος. Δεν είναι ότι δεν ανήκει πια στα κράτη-μέλη. Δεν θα το έλεγα μεταφορά. Είναι 5% που διατίθεται σε αυτό το ε, σκέλος ως εγγύηση για έργα που που θέλει το κράτο μέλο και έχουν εντοπιστεί ω τέτοια, να ε, του εγγυηθεί τη χρηματοδότηση. Αυτό θα βοηθήσει βεβαίω τα κράτη-μέλη που έχουν ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή αναπτυξιακέ τράπεζε πιο αδύναμε. Αυτό διευκολύνει τη χρηματοδότηση. Διότι θα υπάρχει αμέσως πρόσβαση στο τριπλό α και λύνονται και τα προβλήματα των ε, κρατών μελών. Γιατί ο μηχανισμό του InvestEU με τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει και δίνει τι σχετικέ εγγύσει. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρόσθετη δυνατότητα που θα βοηθήσει την εδαφική ισορροπία και τα κράτη-μέλη που είναι λιγότερο ανεπτυγμένα να προχωρήσουν. Είναι μια πρόσθετη ε, διευκόλυνση που οι εμπειρογνώμονε την πρότειναν και ελπίζω ότι και η Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη ε, που συμμετέχει στην εξέταση του θέματο θα το κατανοήσει. Είναι σημαντικό και για τη συνοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χωσέ Μανουέλ. Ζωζέ Μανουέλ. Το λόγο τώρα έχουν οι σκιώδεις ε, Δύο λεπτά έκαστο. παρακαλώ. Ο Παύλο Ρεμπίχ, που ε, αντικαθιστά τον κύριο Κάρας. Ευχαριστώ πολύ,

Δυστυχώ ασθενεί ο κύριο Κάρα, είναι σκιώδης ηγητής του ΕΛΚ στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, στα αγγλικά ο κύριο Ρούμπιχ. Ευχαριστεί του συνεισηγητέ για το σχέδιο έκθεση που είναι γενικά καλή και ισόρροπη βάση για την εργασία των επόμενων εβδομάδων. Καλωσορίζει και χαιρετίζει το σχέδιο έκθεση για να υπάρχει ένα ενιαίο ε, εγχειρίδιο που θα περιγράφονται οι κανόνε σε μία στέγη για όλα τα προγράμματα, καλύτερη πρόσβαση, λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερες επικαλύψεις θα έχουμε. Επίσης, χαιρετίζει την πρόθεση των δύο συνσηγητών να βελτιώσουν την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάζοντας κάποια καλά στοιχεία του ΕΦΣΥ, του Ταμείου Στρατογικών Επενδύσεων, όπως είναι οι πλατφόρμες επενδυτικές, ως συμπληρωματικό προς τις εγγύησεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρή προσθετικότητα για να υπάρχει ψηλή ποιότητα και χρηματοδότηση του ρίσκου όταν υπάρχουν ε, αδυναμίες ε, δανειοδότησης από την αγορά κλπ. Ορισμένες ενισχύσεις επίσης ε, με τη δημιουργία του steering board για πιο καλή διαχείριση και μια ανεξάρτητη επιτροπή διαχείρισης των επενδύσεων με τον έλεγχο και του Κοινοβουλίου με τη διαχείριση του Ταμείου InvestEU και με το συμβουλευτικό κόμβο που θα εξασφαλίζει αποτελεσματική συνεργασία με τους τέρους που εκτελούν τα προγράμματα και την υποστήριξη των μικρομεσαίων και των νεοφυών επιχειρήσεων. Επίσης, 75% της ευρωπαϊκής εγγύησης θα εντράζει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αφού καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα να είναι πολιτικά ανεξάρτητες οι ε, ε, αποφάσεις για τις επενδύσεις και όλα αυτά ρυθμίζονται πολύ καλά, ε, όπως και η μέτρηση του κινδύνου προσοχή μην χαλαρώσει το άρθρο 9 ε, μιλάει για την ε, διατήρηση ε, των σφιχτών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας. Ο εισηγητής προσβλέπει στη συνεργασία και στην καλή απόφαση που θα λάβουμε. Ευχαριστώ κύριε Ρούμπιχ. Να διαβεβάσετε τα περαστικά μας στον κύριο Κάρας. Η κυρία Αίντερ Γαριαθάμπα Ρουμπιάλ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πέντε ιδέες έχω να αναφέρω εγώ. Πρώτον, συμφωνώ με τα όσα έλεγε ο κύριος Φερνάντες και τα έχει γράψει και στην έκθεσή του. Νομίζω θα πρέπει να διατηρήσουμε το επίπεδο της εγγύησης αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στο παρόν PDP ε, για τα χρηματοδοτικά μέσα ε, και τα όσα ίσχυαν για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Το δεύτερο, για τη μεταφορά το 5%. Ξέρω ότι είναι ακαθόδες το θέμα και θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ξέρω ότι είναι μόλις ένα 5% και επίσης γνωρίζω ότι είναι κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών. Αλλά εγώ έχω ένα πρόβλημα αρχής με αυτές τις ιστορίες, γιατί αν πάρουμε χρήματα από την πολιτική συνοχή και τα δίνουμε στις πιο μειονεκτούσες περιοχές, είναι επειδή χρειάζονται χρηματοδότηση ε, ε, για κάποια έργα που μπορούν να γίνουν μόνο με την επιδότηση. Αν βάλουμε τώρα 5% από τα κεφάλαια αυτά σε άλλο ταμείο, που στόχο έχει να καλύψει τις ελλείψεις της αγοράς και δεν έχει καμία σχέση με τα επιδοτούμενα έργα, νομίζω ότι αλλάζει η φιλοσοφία ολόκληρη, έστω και αν είναι 5% η χρηματοδότηση. Το πιο λογικό πάντως θα ήταν να συζητήσουμε με τους συναδέλφους Επιτροπής Ρέτζι για να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε αυτό με ασφαλιστικές δικλίδες. Τρίτον, προφανώς και μια που μιλάμε για το ΕΦΣΙ, θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με προσθετικότητα. Βελτιώσαμε από το ΕΦΣΙ 1 στο ΕΦΣΙ 2, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια έργα που μπορεί να δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες, αν θα πρέπει πραγματικά να χρηματοδοτούνται από αυτόν τον μηχανισμό και ούτε μπορούμε να κάνουμε ανταγωνισμό σε άλλες αναπτυξιακές εθνικές τράπεζες που ήδη ε, λειτουργούν στην αγορά. Αυτό θα πρέπει να είναι έτσι μια πρόσθεση και όχι ε, υποκατάστατο. Το τέταρτο έχει να κάνει με τη διαχείριση. υπήρχε κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Γι' αυτό έχουμε καταργήσει το προηγούμενο σύστημα, αλλά θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χάσουμε το ελεγκτικό όργανο που αξιολογεί και τα έργα. Και το πέμπτο, για το InvestEU, θα πρέπει να ε, μιλούν εκεί και ειδικοί για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ε, θέματα. Ο κύριος Λούνας. Ευχαριστώ. Αύριο ξεκινάμε. Αύριο θα εμφανιστεί ο δείκτης ε, των διευθυντών επιχειρήσεων, ε, των υπευθύνων αγορών, κάτι το οποίο μας δείχνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αρχίζει να επιβραδύνει και ε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε το επενδυτικό κλίμα γιατί πρέπει να κάνουμε περισσότερα, οπότε καλώς ορίζω αυτήν την πρόταση. Ας δούμε λοιπόν το επενδυτικό κλίμα Ας δούμε τα νομοθετικά εμπόδια, ίσως είναι ακόμα υπερβολικά και ίσως είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια. Ας δούμε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, υπάρχουν πολλά που πρέπει να επιληθούν, ας δούμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά ας δούμε και αυτό το θέμα, το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε επενδυτικέ ευκαιρίες σε ένα εργαλείο. Κοιτώντας λοιπόν την πρόταση της Κομισιόν, νομίζω ότι είναι λογικό να απλοποιήσουμε το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα 14 δηλαδή χρηματοδοτικά μέσα να ε, ενωθούν και είμαστε έτοιμοι ακριβώς ε, να συνεργαστούμε επικοδομητικά και γρήγορα. Αλλά διαβάζοντας εδώ την πρόταση της Κομισιόν έχω και κάποιες ερωτήσεις ειδικά για την σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ήταν νομίζω λάθος το να μην συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην σύνταξη αυτή τη ε, έκθεση. Ε, ίσως να είναι ζήτημα σχέσεων μεταξύ τη Τράπεζα Επενδύσεων και τη ε, Κομισιόν. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να συμφιλειωθούν αυτά τα δύο θεσμικά όργανα και αυτό θα γίνει μέσω του σεβασμού των αρμοδιοτήτων του καθενό και των ευθυνών του. Και έρχομαι έτσι στην διακυβέρνηση του έργου την διοίκησή του. Ίσως να είναι λίγο νωρίς γιατί Κομισιόν είχε στόχο να αποκτήσει τραπεζική πείρα, ενώ για εμάς ο φυσικός εταίρο τη Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα τραπεζικά καθήκοντα και η πρόταση των εισηγητών πάει σε μια πιο λογική κατεύθυνση, δηλαδή ο καθένα έχει διακριτού. ρόλους. Τώρα, για το λεγόμενο συνικό τείχο που θα το διαχωρίζει, εντάξει, καλέ ιδέε. και επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, θα ήθελα να τονίσω τον ρόλο των εθνικών ε, τέτοιων τραπεζών που έχουν ένα ρόλο να παίξουν για να επιτυχημένο αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ, Μπεν ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τους εισηγητές για την δουλειά που έκαναν και επί της αρχής νομίζω δεν έχει κανείς καμία αντίρρηση, είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση Προσπαθούμε δηλαδή να συνενώσουμε, να εναρμονίσουμε διαφορετικά προγράμματα για να μειωθεί και το διοικητικό βάρος και για τον χρήστη και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Βεβαίως πρέπει να ομολογήσω πως εγώ έχω διαφορετική άποψη από όσες ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι επιτυχημένο. Το ακούμε συνεχώς να λέγεται, αλλά εγώ δεν έχω συγκεκριμένα δεδομένα για κάτι τέτοιο, ειδικά όσον αφορά την προσθετικότητα, κάτι το οποίο καθόλου δεν αποδεικνύει την επιτυχία του ΕΦΣΙ, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Μπορεί ο στόχος να είναι να διαθέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει να είναι επιπρόσθετα, που δεν θα υπήρχαν δηλαδή, χωρίς αυτό το ταμείο και να είναι βιώσιμα, κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχθεί. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για πράγματα τα οποία θα θέλαμε να έχουμε, αλλά δεν υπάρχουν. Επιπλέον, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όλα τα χρηματοδοτικά μέσα είναι αυτό το οποίο λέει το όνομα. Χρηματοδοτικά μέσα, δηλαδή χρηματοδοτούνται εδώ πέρα προγράμματα, κάτι το οποίο σημαίνει πιστώσεις. Μπορούμε να βγάλουμε 100 διάφορα ωραία ονόματα, αλλά φοβάμαι ότι ε, θα δούμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις που είχαμε πριν από 10 χρόνια και τότε είχαμε κάποια χρηματοδοτικά μέσα όπου ήταν πάρα πολύ ωραία αλλά κανείς δεν τα καταλάβαινε και οδηγήθηκαμε σε μια τραπεζική κρίση η οποία εκτροχίασε την παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως αυτό δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στην παγκόσμια οικονομία αλλά είναι ένα τμήμα του το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι απλούστερο. Υπάρχουν λεφτά στις ε, αγορές, έχουμε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί τα κάνουμε τα πράγματα τόσο δύσκολα και περίπλοκα. Θα ήταν λογικότερο και ουσιαστικότερο να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική συνοχή και βεβαίω να προωθήσουμε τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, είναι η αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξουμε, αλλά όχι κάποια προγράμματα στα οποία ε, κανείς δεν ξέρει τελικά και τι σημαίνουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύντομα, γιατί έχουμε δύο λεπτά μόνο ο καθένας. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν προηγουμένως. Για να πω κάτι καινούριο, έχει έρθει η ώρα να ενισχύσουμε ε, ε, την απόδοση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, δηλαδή να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα με ανάπτυξη του ΑΕΠ και με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Σε κάποια κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να φτάνουν επιτέλους ε, στις σωστές ε, επιχειρήσεις αυτά τα χρήματα που είναι στραμμένες προς την πράσινη οικονομία, προς την καινοτομία και να μην έχουμε το τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα, ε, καταλήγουν στις τσέπες κάποιων ολιγαρχών για να κάνουν ό,τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε τα ομόλογα έργου και στην, στην ε, Ισπανία ε, αυτά τα ομόλογα εργού κατέληξαν στις τσέπες εκείνων που ε, σχεδίασαν ένα μεγάλο έργο ενεργειακό που προκαλεί σεισμούς στις ακτές της χώρας. δεν θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευκαιρία των αγορών το πώς θα μοιράζουν αυτά τα χρήματα, να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και μεγέθυνση της οικονομίας. Και ως ε, φιλελεύθερος από τη Μεσόγειο θέλω να σας πω ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε μία τεράστια Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιανομής με μεταφορά πιστώσεων από το βορρά στο νότο, αλλά να εναρμονίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, να πηγαίνουν σωστά τα χρήματα στους σωστούς δικαιώους. Αυτά θέλουμε, όχι μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο λεπτά ακριβώς. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Ε, ο κύριος Τόρβαλς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ζωζέ Μανουέλ και τον Ρομπέρτο για την πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει. Εχθές στη συνεδρίαση των σκιωδών μας υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουν μια εικόνα, ένα διάγραμμα για το πώς φαντάζονται τη διακυβέρνηση. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για πολλούς λόγους, μερικούς από τους οποίους ακούσαμε σήμερα στη συζήτηση. Γιατί θα γίνει μεγάλο παζάρι ε, γύρω από το πώς θα γίνει η διακυβέρνηση και θέλουμε να δούμε πού θα ε, κατασταλάξουν όλα αυτά. Επίσης θέλουμε να δούμε το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνική βιωσιμότητα να εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές και αποδεδειγμένα. Και εδώ τίθεται το εξής νέο ερώτημα. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος για να τα αποδείξουμε όλα αυτά. Γιατί δημιουργήσαμε κάτι πολύ γραφειοκρατικό και δεν χρειάζεται τέτοια γραφειοκρατία. Πού θα γίνονται οι έλεγχοι και πώς θα γίνονται με εύκολο τρόπο σε αυτή τη δομή διακυβέρνησης. Μετά, η δυνατότητα εθελοντικής ε, χρησιμοποίησης κονδυλίων από τη συνοχή, είτε ως συνεισφορά, είτε ως μεταφορέ. Οι φιλελεύθεροι ε, που είναι στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν άλλη άποψη, θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, έχω και κάποιες ερωτήσεις. Για ποιο λόγο προτιμάμε τον ορισμό του FC2 για την προσθετικότητα σε σχέση με αυτό που υπάρχει ε, στον δημοσιονομικό κανονισμό. Γιατί χρησιμοποιείται αυτό τον ορισμό. Και μετά έχουμε διάφορα πολιτιστικά και δημιουργικά σε αυτό το φάκελο και καμιά φορά εγώ έχω πρόβλημα με τον ορισμό το ίδιο. Τι εστί δημιουργικότητα και τι εστί πολιτισμός. Αν δεν βάλουμε κάποια όρια εκεί, νομίζω θα μεταφραστεί ως ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και επίσης τα διάφορα όργανα, τα διοικητικά, ε, έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα ή όχι. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Σβέν Γκίγκολτ. Απόν. Ο Γιώργη Σολέ, λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος και του συναδέλφου Σπεν Γκίγκολ, ο οποίος ασθενεί και αυτός δυστυχώς. Ε, γενικά συμφωνούμε με την ιδέα να συνενωθούν ε, ε, τα πολλαπλά χρηματοδοτικά μέσα που υπάρχουν σήμερα. Καλό είναι αυτό. Αλλά τώρα η δουλειά μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις που υποστηρίζονται από το μέσο αυτό να είναι οι καταλληλότερες για μια βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια αυτή, ο βασικός στόχος ε, που ε, επιδιώκουμε και μέσω των τροπολογιών μας είναι το InvestEU, να παραμείνει ευθυγραμμισμένο με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς στόχους για το κλίμα. Μεταξύ αυτών, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι τομεί πολιτικής θα πρέπει να ελέγχονται από την πλευρά της ε, ε, βιωσιμότητας και να παρακολουθούνται και της κοινωνικής, της περιβαλλοντικής και λοιπής για να ε, περιορίζονται όσο γίνεται επιβλαβείς επιπτώσεις και να ενισχύεται η θετική του συνεισφορά. Και μια κατεξουδότηση πράξη θα για ένα πλαίσιο εξασφάλισης βιώσιμης επένδυσης. Για να ελέγχουμε κάθε φορά αν μια οικονομική δραστηριότητα είναι βιώσιμη με βάση τους στόχους για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, επίσης, ακούστηκε και μια ιδέα με την οποία συμφωνούμε στην Επιτροπή ε, Ήτρε Βιομηχανίας να έχουμε μια νέα θηρίδα για την ανακαίνιση κτηρίων όπου να χρηματοδοτούνται ε, και ιδιώτες ε, και συλλογικότητες με επενδυτικέ πλατφόρμες για την ανακαίνιση των κτηρίων με φορολογικές ελαφρύσεις. Κατά την άποψή μας, το είπα και χτες, στη συνεδρία των Σκιωδών, το δεύτερο παράρτημα χρειάζεται αναθεώρηση και να είναι μια, ένας αποκλειστικός κατάλογος, εξαντλητικός κατάλογος των ε, δραστηριοτήτων που καλύπτονται και θα κάνουμε και προτάσεις για ξεχωριστά άρθρα καινούρια σε σχέση με αυτό και θα κάνουμε και προτάσεις για να αυξηθεί η λογοδοσία και η διαφάνεια ε, των δομών διακυβέρνησης και να είναι και πιο στιβαρό το βαθμολόγιο. Ευχαριστώ κύριε Σολέ. Πείτε και εσείς περαστικά στο Σφεν Κίγκολτ από πλευρά μας. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης παρακαλώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές. Ε, θεωρώ το κείμενο για το InvestEU μια καλή βάση για το διάλογο που διεξάγουμε. Αποτελεί ουσιαστικά μια εμπλουτισμένη συνέχεια της εμπειρίας που έχουμε από το EFSI, το γνωστό ως Ταμείο Γιούνκερ. Ο στόχος νομίζω ε, αυτού του νέου εργαλείου, αυτής της νέας δομής είναι να αντιμετωπίσουμε τα επενδυτικά κενά που υπάρχουν και συνεχίζονται ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αμβλύνουμε τις ε, ανισότητες ανάμεσα σε κράτη-μέλη και σε περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει ακόμη πιο έντονα και συνδυαστικά με τις πολιτικές συνοχής να αντιμετωπίσουμε περιφερειακές ανισότητες, ιδιαίτερα με στήριξη περιοχών όπου υπάρχει υψηλή αποεπένδυση και υψηλή μακροχρόνια ανεργία. Θα θέλαμε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο. Φυσικά αυτό συνδυάζεται και με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είναι δυστυχώς ακόμη σε εκκρεμότητα για να ενισχύσουμε βιώσιμες περιβαλλοντικές υποδομές, την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την κοινωνική οικονομία, περισσότερες ευκαιρίες για την νεολαία, ενίσχυση της ψηφιακής σύνδεσης, πιο αποτελεσματικές μεταφορές, ενίσχυση της πράσινης καινοτομίας και της κοινωνικής οικονομίας. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την δυνατότητα συμμετοχής και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και μιλώντας για τα τέσσερα παράθυρα που προβλέπει ε, η πρόταση, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της κοινωνικής επένδυσης. Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντικό και προτείνω να ενισχυθεί το ρόλο του Advisory Hub για τις χώρες που είχαν και πέρασαν μια μεγάλη κρίση γιατί εκεί υπάρχουν σημαντικά μικρής κλίμακας προγράμματα που θα πρέπει να ενισχυθούν. Στην ε, επόμενη φάση θα καταθέσουμε προτάσεις σε συνεργασία με τους συζητητές και τους άλλους κοιόδης συζητητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ εκ μέρου τη ομάδα μου, τη ΕΝΕΦ, και εκ μέρου του σκιώδου εισηγητή που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, στο πρόγραμμα μα. Ε, βλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους στόχους, διότι το κενό των επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη είναι κάτι το προφανές. Και τα τελευταία 8 χρόνια με την κρίση έχει ενταθεί. Οι επενδύσεις και η σόρευση κεφαλαίου για τις υποδομές έχει μειωθεί. Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον αυτό το εργαλείο θα είναι αποτελεσματικό και θα δώσει ένα σπρόξιμο, μια ορμή ε, μια νέα ορμή στι επενδύσει, κάτι που τόσο χρειάζονται. Ε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πολλέ απόπειρε να τονώσουν, να παρακινήσουν και να υποδαβλήσουν τι επενδύσει, ιδίω στι υποδομέ, με διάφορα εργαλεία και διάφορου μηχανισμού. Ξεκινήσαμε το 2011 με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με το Project Bond Initiative, την πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η χρηματοοικονομική ε, δομή για να δοθεί κίνητρο για μεγάλα διακρατικά έργα. Τώρα υπάρχει το πρόγραμμα Juncker και προσπαθούμε στον προπολογισμό να προβλέψουμε πλέον ένα εργαλείο τέτοια φύση, τέτοιων διαστάσεων. Ε, είναι σαφές ότι για να λειτουργήσει το εργαλείο αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερο τη χρήση. Δηλαδή και ως προς την φάση επιλογής των έργων μέχρι τη φάση της υλοποίησης, αλλά και ως προς τους όρους λειτουργίας της εγγύησης και εδώ τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν πρέπει να είναι κριτήρια που και η αγορά και οι φορείς της αγοράς να μπορούν να δεχτούν ώστε να γίνουν αυτές οι επενδύσεις και για τους ε, ε, δικαιούχου των επενδύσεων από αυτού που θα λάβουν τι επενδύσει. Χωρί αυτά τα δύο σκέλη, δεν βλέπω στην πραγματική υλοποίηση να τα καταφέρουμε, να δοθεί αυτό το ε, αυτή η απαραίτητη όθηση στι επενδύσει που θέλουμε να δώσουμε για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκτό των σκιωδών εισηγητών, υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Ένα λεπτό. Για όποιον τον θέλει. Καλημέρα σας. Ε, επειδή είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής αν μπορείτε. Το πρόγραμμα Juncker, το ΕΦΣΙ, όταν επινοήθηκε, Υποτίθεται ότι ήταν ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τις, ε, τα μη προβλέψιμα στοιχεία των οικονομικών κύκλων. Δηλαδή κάτι που θα έπρεπε να καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για σταθεροποίηση. Το ε, εργαλείο που συζητάμε όμω τώρα είναι σαν να έρχεται να συμπληρώσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι νέα τράπεζα επενδύσεων, είναι ένας προπολογισμός ε, μέρος δεύτερο, κάτι το συμπληρωματικό, σε περίπτωση το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στο το προηγούμενο. Θα καταφέρουμε λοιπόν να λειτουργήσει μοχλευτικά αυτό το εργαλείο για να αποφύγουμε του κλειδονισμού των διάφορων ε, αλλαγών στους οικονομικού κύκλου. Ε, Πρόεδρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να απαντήσει. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, λίγα λόγια από την πλευρά μα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του δύο συνεισηγητέ για την ε, πολύ καλά προετοιμασμένη εκθέσή του, Πραγματικά έχει επικεντρωθεί στην ουσία τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. την ανάγκη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τι επενδύσει. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει όπου τα κενά των επενδύσεων καλύπτονται, αλλά σε άλλα κομμάτια τη αγορά υπάρχουν ακόμα πιέσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εδώ λοιπόν σημαντικό είναι να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη ζήτηση και τη φύσης των χρηματοδοτικών εργαλείων και του πολιτικού χαρακτήρα αυτή της πρωτοβουλίας του InvestEU. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε και εκεί το Κοινοβούλιο μπορεί να τονίσει το σκέλος της διαφάνειας και της λογοδοσίας με τις προτάσεις του επικοδομητικά. Καλωσορίζω την έμφαση που δίνεται στην βιωσιμότητα, την κοινωνική και περιβαλλοντική συνοχή. Δεν είναι μόνο θέμα του χρηματοδοτικού εργαλείου αυτού, αλλά εδώ είναι πολύ σημαντικό το σκέλος της συμμετοχής των κρατών μελών. Επίσης, πολύ σημαντική είναι, σημαντική είναι η προστατικότητα. Ε, Καλωσορίζουμε λοιπόν τις προτάσεις του Κοινοβουλίου σχετικά και βεβαίως υπάρχουν τομείς όπου θα θέλαμε να έχουμε στενότερη συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να βρούμε λύσεις. Τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση και μερικά στοιχεία του σκέλους που αφορά τα κρατημέλη. Με αυτά τα σχόλια και αν υπάρχουν ερωτήσεις, κάποια στοιχεία του σκέλους των κρατών μελών ήταν το τελευταίο που είπα. Très bien. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε, θα δώσουμε το λόγο στους δύο συνεισηγητές μας. Τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ο Ζωζέ Μανουέλ θα ξεκινήσει. Αποφασίστε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι, να ξεκινήσω. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Το πρώτο. Το θέμα του σκέλους της συνεισφοράς των κατοβελών. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει διστακτικότητα εδώ. Υπάρχει φόβος. Όμως πρέπει τα κράτη-μέλη να σκεφτούν ότι μπορούν σε αυτό το σκέλος, με την πρόταση που έχουμε τώρα 5%, να ε, προσφέρουν για να προστατεύσουν χώρες με αδύναμες ε, οικονομικές αγορές και έτσι να προασπιστούν και την πολιτική συνοχή. Δηλαδή, αυτοί που είναι προασπιστές της πολιτικής συνοχής, ουσιαστικά ζημιώνουν τις χώρες τη πολιτική συνοχή μεταξύ των οποίων της Πορτογαλία που είναι ένα καλό παράδειγμα. Ε, η πολιτική συνοχή τα χρηματοδοτεί όλα ω προ τις δαπάνε Στη χώρα μου, όχι υποδομές όμως. Στην Πορτογαλία, οι κοινωνικοί θεσμοί, οι κοινωνικοί φορεί χρεώνονται, πάνε στην τράπεζα για να φτιάξουν υποδομές, ε, γιατί οι σχέσεις ε, συνεταιριστικές με, τις, ε, με τα, με τα κονδύλια συνεχής, αυτά μπορούν να πάρουν τα κονδύλια συνεχής, δεν το επιτρέπουν. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει συμπλήρωμα, συμπληρωματικότητα. Είναι μια μορφή και τι λέει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν υποβάλλεται μια πρόταση για, μια, για ένα συνεταιρισμό, ε, έχουμε την εγγύηση του 5%. Δεν θα χρειαστεί σε πρώτη φάση. Όμως ένα μεταγενέστερο στάδιο αυτή τη σύμβαση που βασίζεται σε συνεργασία, μπορεί το κράτο μέλο να χρειαστεί να πάει σε αυτή τη θηρίδα ε, και να μην υπάρξει άλλη ανάγκη. Εδώ λοιπόν είναι κάτι που προβλέπεται για την περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή, αναθεώρηση στι συμβάσει αυτέ. Τα κράτη-μέλη ε, παίρνουν ένα μέρο ε, των διαφορετικών κονδυλίων για την εγγύηση και ουσιαστικά δίνουν την εγγύηση για μεγαλύτερο διάστημα από το που Για την Πορτογαλία, α πούμε, για την οποία μιλάμε. Το 5% του χρηματοδοτικού αυτού ε, χαρτοφυλακίου μπορεί να κινητοποιήσει πάνω από 50.000 ευρώ. Δηλαδή το διπλάσιο από την πολιτική τη συνοχή. Άρα, ξέρουμε ότι η πολιτική συνοχή έχει και τα όρια τη. Εάν έρθουν έργα και προγράμματα ε, υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα αν έρθουν να προσθεθούν από αυτό το παράθυρο, δημιουργούμε σχέσει συνεργασία και έργα που είναι ζωτική σημασία για τα κράτη-μέλη δεν εμποδίζονται. Γιατί να το μπλοκάρουμε αυτό, γιατί να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τις και συμφωνώ ότι ναι, καλό είναι να ενισχύσουμε την προσθετικότητα. Έχουμε προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση για το θέμα της διακυβέρνησης. Θέλουμε ιδέες για να δούμε πώς θα γίνεται σωστά η αξιολόγηση και η επιλογή των έργων. Υπάρχει και άλλη μια δυνατότητα. Υπάρχει και το πρόγραμμα Juncker για την Αφρική. Εκεί είναι παρόμοια η φιλοσοφία που έχει εφαρμοστεί. Δηλαδή θα υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι είτε θα αξιολογούν, θα κάνουν το assessment των έργων από το του InvestEU και μετά και των έργων που υποβάλλονται στα πλαίσια του προγράμματος Juncker για την Αφρική. Αυτή τη στιγμή είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει αυτή την ονομασία. Αλλά εδώ θέλουμε και περιορισμό του γραφειοκρατικού άκθου. Να αποφύγουμε τι συγκρούσει συμφερόντων. Είναι και αυτό ζωτική σημασία. Είναι από του λόγου για του οποίου το πρόγραμμα team δεν το προτιμήσαμε. Η ειδική μια εθνική ε, ειδική τράπεζα δεν μπορεί να αξιολογούν προγράμματα των ανταγωνιστών του. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Δεν είναι λογικό. Και για την προβλεψιμότητα και αυτό το 25% για τους άλλους εταίρους ε, που θα είναι implementing partners έχει λογική. Νομίζω ότι επιτρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα που όλοι απαιτούν. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και όταν πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει φούσκα στα ακίνητα, πληθωρισμό. Εδώ σκέφτομαι στη Λισαβόνα πόσο έχει ανέβει το τετραγωνικό. Για άλλους λόγους λέει ο κ. δεν φταίει αυτό. Δεν είναι από την πολλή ανάπτυξη. Και τώρα το λόγο έχει ο Ρομπέρτο Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και ηγητές για την θετική προσέγγιση και τις επικοδομητικές συνεισφορές τους. Και αναμένουμε τις τροπολογίες τους για να συζητήσουμε πιθανές ε, λύσεις ε, και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις με βάση την συζήτηση για τα εθνικά αυτά τμήματα. Πράγματι προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες δικλίδες ασφαλείας. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν συμφωνώ τόσο το ότι εξορισμού ένα τέτοιο μέσο δεν είναι συμβατό με την φιλοσοφία της πολιτικής συνοχής. Πρώτα απ' όλα, αν ε, δεν κάνω λάθος, υπάρχει η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή και τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο. Ε, είναι ένα άλλο όνομα, ένας άλλος τρόπος να κάνουμε κάτι το οποίο είναι ήδη δυνατό. Και έτσι μπορούμε να έχουμε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά μεταξύ των οποίων και η ανάμειξη χρηματοδοτικών μέσων με το άλλα τμήματα του Ταμείου Συνοχής. Οπότε αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο εάν το δούμε σωστά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα μας δώσει την δυνατότητα ε, να έχουμε κάποια εργαλεία για τους ε, στόχους του Ταμείου Συνοχής, ε, το οποίο έχει τους στόχους, δεν ξεχνάμε. Οπότε έχουμε ήδη πολλούς τομείς που αλληλεπικαλύπτονται γι' αυτό ακριβώς. Έχουμε τα διαφορά χρηματοδοτικά μέσα σε περιφερειακό επίπεδο Και βεβαίω ε, υπάρχουν κάποιε βελτιώσει. Θα συζητήσουμε με του συναδέλφου τη Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων, αλλά δεν συμφωνώ ότι είναι ασύμβατο. Ε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, θα πρέπει να μην. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ αφενός ε, του να βασιστούμε στην πείρα του ΕΦΣΥ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να έχουν μεγαλύτερο ρόλο οι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Υπάρχει νομίζω αυτή η ισορροπία στο κείμενο, μπορεί να βελτιωθεί, αλλά και από την συζήτηση που ακούσαμε κάπου εκεί βρισκόμαστε. Ο κύριος Τόρβαλτς έκανε μια καλή ερώτηση γιατί ελαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις του κυρίου Τρεμόζα πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, διάσταση της ε, ποιότητα που πρέπει να βελτιωθεί. Ε, διαφωνώ με του που λένε ότι το FC δεν ήταν επιτυχία. Ήταν τεράστια επιτυχία, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Οπότε υπό μία έννοια το σκεπτικό εδώ πέρα είναι ότι έχουμε τον εταίρο ο οποίος κάνει μία πρόταση έργου, μετά η Κομισιόν ελέγχει το εάν αυτά συμφωνούν ε, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Μετά γίνεται η αξιολόγηση από τον εφαρμοστικό εταίρο με βάση μια βαθμολογία. Ξανά έλεγχο από την Κομισιόν και μετά πάει στην Επενδυτική Επιτροπή. Δηλαδή ακόμα και με αυτό το νέο σύστημα, Χωρί την ομάδα έργου, ε, υπάρχουν ε, φάσεις στην διαδικασία όσον αφορά και τον πίνακα της βαθμολογίας και τους ελέγχους που θα διασφαλίσουν ότι η ποιότητα και η διάσταση της πολιτικής δεν ε, χάνεται και δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε τα χρήματα σε κάποιους εταίρους εγγυημένα και θα τα κάνουν ό,τι θέλουν. Από την άλλη βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο ευελιξίας, ε, προσαρμογής, αλλιώς κινδυνεύουμε να μην υπάρχει δυνατότητα να έχει αποτελέσματα. Να μην έχουμε δηλαδή έναν πολύ γραφειοκρατικό και δίσκαμπτο μηχανισμό. Έχουμε βρει λοιπόν μια ισορροπία, μπορούμε να δουλέψουμε, να ακούσουμε σχόλια. Αυτή ήταν όμως η φιλοσοφία, το σκεπτικό των τροπολογιών μας. Τέλος, να διαβεβαιώσω τον κύριο Κάρας ε, και τον συνάδελφο που τον εκπροσώπησε ότι υπάρχει αυτή η διάταξη των μέτρων άπαξ, κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στο ΕΨΙ για τις εθνικές πλατφόρμες. Μπορούμε λοιπόν να το βελτιώσουμε αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι κάποιο τεράστιο εμπόδιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τους δύο. Α, θέλετε το λόγο. Διαδικαστικό, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Λόνας. Πολύ σύντομα. Ακούω μεγάλη προθυμία να εργαστούμε γι' αυτό, γιατί τι μελλοντικέ συνεδριάσεις ενδεχομένως να ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και τη λέει Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τώρα μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούσαμε. Μάλιστα, το σημειώσαμε. Ε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και τους δύο συνεισηγητές. Ε, νομίζω ότι πάει καλά το πράγμα και είναι πολύ μεγάλη η συνένεση. Ας ελπίσουμε να μην τσακωθεί τώρα η Κομισιόν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν αμφιβάλλω ότι θα επηρεάσει και τις επενδύσεις ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η διακυβέρνηση αυτών των συστημάτων. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 6 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε μαζί στις 3 Δεκεμβρίου σε κοινή συνεδρίαση. Τούτων όλων λεχθέντων κλείνει εδώ το πρώτο μέρος και δίνω το λόγο στον Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη που θα προεδρεύσει το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης. Ευχαριστώ, Ζα. Ας περάσουμε σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα και επίκαιρο, το οποίο είναι, και γιατί δεν το βρίσκω αφού είναι τόσο σημαντικό. Just a second. Somewhere. Κάπου το έχω. Uh, uh, Ωραία, το βρήκαμε. Ε, ε, Δημιουργία ενός μηχανισμού για τη σταθεροποίηση ε, που είναι βασικό στοιχείο στη συζήτηση για την ολοκλήρωση και βάθηση της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, Δύο εισηγητές έχουμε ε, και εδώ. Όπως ξέρετε έχουν εργαστεί στις εκθέσεις τους, τις έχουν εκπονήσει και κατέθεσαν ένα κείμενο. Και θα δώσω το λόγο στους δύο εισηγητές μας, ε, πέντε λεπτά ο καθένας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αρχίσει, ο Ράιμερ Μπέγκε. ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι Κομισιόν κατά αυτήν την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθεροποίησης και Επενδύσεων είναι ενσωματωμένη στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αφετός ε, μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση αυτή από μόνη τη. Ε, βγάζει τα απαραίτητα συμπεράσματα από την εμπειρία της διαχείρισης των κρίσεων ε, και των διεθνών αγορών. Από την άλλη θεωρώ ότι είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο να δούμε το συνολικό πλαίσιο της ε, στρατηγικής ε, τοποθέτησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ΠΔΠ. Βεβαίως τα πακέτα αυτά κάπου πάνε μαζί, τα νέα μέσα τα οποία συζητήσαμε την Δευτέρα και σήμερα, αλλά και το ερώτημα του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αδυναμίες στα μεγάλα ταμεία μας όσον αφορά την αηφορία, όσον αφορά τις ε, προσδοκίες προώθησης ε, της ανάπτυξης, ε, της απασχόλησης, να καταπολεμήσουμε την ανεργία και ποια αιρεσιμότητα θα πρέπει να υπάρχει για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε και την τάξη μεγέθυνση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Αυτά νομίζω πάνε μαζί για να βρούμε μια αξιόπιστη απάντηση. Δεύτερη παρατήρηση επανέρχομαι λίγο σε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε την ε, έκθεση Δίας πρωτοβουλίας του Φεβρουαρίου 2007 η οποία τελικά βεβαίω πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία για την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Ο τίτλος σήμερα βεβαίως είναι διαφορετικός αλλά το περιεχόμενο έχει μεγάλη σχέση. Και με βάση τα όσα αποφάσισε η Ολομέλεια για τα θέματα των ασύμετρων κραδασμών και σόκο, τα οποία βεβαίως δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν και αν θα έρθουν, αλλά ένα μάθημα το οποίο αντλήσαμε είτε μιλάμε για την προσφυγική κρίση είτε για την τραπεζική κρίση είναι ότι στο παρελθόν δεν ασχοληθήκαν ποτέ προληπτικά με την διαχείριση κρίσεων και αυτό το απαιτούν από μας οι πολίτες. Έχουμε λοιπόν ε, ζητάμε εδώ πέρα ξεκάθαρους κανόνες για έναν αυτόματο μηχανισμό απορρόφησης κραδασμών, σαφείς κανόνες ποιος πληρώνει, ποιος λαμβάνει, υπό ποιες συνθήκες και με ποιον τρόπο και πώς θα είναι αυτό μακροπρόθεσμα ουδέτερο δημοσιονομικά όπως λέγεται. Έχουμε συζητήσει επίσης για την μορφή της ε, διακυβέρνησης και εάν δούμε την πρόταση Κομισιόν υπ' αυτό το πρίσμα, είναι μια προσεκτική πρόταση. Αν δείτε τα εκτιμώντας ε, όσον αφορά την εξέλιξη αυτής της ιδέας ε, του Ταμείου Σταθεροποίησης και Επενδύσεων, πάρα πολύ συχνά λέει θα μπορούσαμε, θα έπρεπε, ε, θέμε ή δεν θέμε τελικά. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω πω υπάρχει και ένα διχασμό εντό του Συμβουλίου. Τα μισά κρατημέλη είναι υπέρ τη πρόταση και ένα τμήμα 14-15 ε, κρατών μελών είναι ανοιχτό σε μια συζήτηση. Αλλά βεβαίω γύρεται το ερώτημα του ηθικού κινδύνου κτλ. Ε, πριν μπορέσει να συμφωνήσει με την άλλη πλευρά. Οπότε πρέπει εδώ πέρα να γίνει ένας απολογισμός και θα έλεγα ότι κατά την απόψή μας το θέμα δεν να πούμε ναι ή όχι, αλλά α, πότε και πώς και ποιος. Και αν δούμε τώρα κάποιες ε, προτάσεις που υπάρχουν ε, στην ε, πρόταση της Κομισιόν, θα φέρουμε βεβαίω και κάποιες ε, διορθωτικές ε, προτάσεις, δηλαδή το 30 δισεκατομμύρια το ποσό που προβλέπετε είναι 0,3% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Και με τέτοια ποσά ίσως να αντιμετωπιστούν ε, τα σοκ μικρότερων χωρών, αλλά όχι των μεγαλύτερων, οι ασύμετροι κράτασμοι. Δεύτερον, οι ειδικοί με τους οποίους το συζητήσαμε εντατικά Είπαμε ότι το κριτήριο ενεργοποίησης είναι κάτι το λογικό, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας αυτοματισμός με ξεκάθαρες συνθήκες που θα ενεργοποιηθεί, με ξεκάθαρες συνθήκες και να μην ρεζιλευόμαστε με συζητήσεις που θα καρτάνε μήνες. Οπότε, με το μηχανισμό ενεργοποίησης και με την έννοια αυτή της τάξης μεγέθους θα μπορούσαμε ίσως να διαπραγματευτούμε λογικά για ένα τέτοιο μέσο και να υπάρχει μια σταθεροποίηση των ε, επενδύσεων ε, και μέσω του ESM. Και βεβαίως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε να μην χάσουν οι χώρες επενδύσεις οι οποίες προετοιμάζονται έτσι μέσω ε, να μην τις χάσουμε μέσω αυτού του μηχανισμού. Αν δούμε λοιπόν το θέμα των εισφορών. Έχουμε την έκθεση ίδιας ε, πρωτοβουλίας, έχουμε μιλήσει για εισφορές των κρατών μελών με βάση τα έσοδα, έχουμε επίσης ε, το μέσο του ισοζυγίου πληρωμών, υπάρχει εκεί πέρα ακουστή το νούμερο των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν πολλέ ε, δυνατότητε. Κάποιοι μίλησαν για ένα τμήμα των κερδών της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας ε, για να συνδεθεί με, και με τη λειτουργία της Ευρωζώνης. Αλλά θα πρέπει βεβαίως να είναι αξιόπιστες οι προτάσεις. Ταυτόχρονα είναι σαφές. Και αυτό δεν είναι απλά η ιδέα δύο εισηγητών από δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες ότι σε βάθο χρόνου χρειαζόμαστε ένα σύστημα ασφάλισης ε, γιατί βεβαίως ένα σύστημα αντασφάλισης ε, πληρώνει κανείς, ε, πληρεί τις συνθήκες και αναλόγως κινείται. Και αυτό το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Κλάου Ρέγκλινγκ γιατί λέει ότι οι αγορές περιμένουν ένα τέτοιο μέσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και πολλοί διάφοροι επιστήμονες από διαφορετικές οικονομικές σχολές είχαν τοποθετηθεί υπέρ ε, κάποιου τέτοιου συστήματος και βεβαίω ε, το ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ ε, δεν πρέπει μόνο να το καλούμε για κάποιες χώρες που έχουν περάσει σε κρίση και μετά όταν μας λέει χρειάζεται κάτι τέτοιο να μην το ακούμε. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Να λοιπόν που επανερχόμαστε ε, στη συνέχεια, την άμεση συνέχεια της προηγούμενης έκθεσης που συνεκπονήσαμε με το Ράιμερ Burger, ε, σε ένα διαφορετικό όμως πλαίσιο σήμερα. Ο λόγος ύπαρξης ε, του μέσου αυτού που θα συζητήσουμε ε, γίνεται επιτακτικότερος μέρα με τη μέρα. Γιατί όλοι συνειδητοποιούν ότι αν δεν υπάρχει αυτόματο σταθεροποιητής, όπως το είπαμε και στην προηγούμενη έκθεσή μας, η Ευρωζώνη θα μπορούσε να γνωρίσει κρίσιμους κραδασμούς. Ε, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα μέσο και ο λόγο ύπαρξη είναι ένα από του πυλώνε που είχαμε εντοπίσει και στη δική μα έκθεση ενό ασύμετρου κραδασμού. Είδαμε τι γίνεται και με του συμμετρικούς κραδασμού και με τη σύγκληση, αλλά αυτό δεν πρόκειται για το ε, για τους συμμετρικούς αλλά για τους ασύμετρους κραδασμούς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το δεύτερο είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να είναι αυτόματος αυτός ο σταθεροποιητής. Αυτός θα πρέπει να είναι λοιπόν ο ερμός της σκέψης μας. Και με βάση αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα κριτήριο ενεργοποίησης του αυτόματου σταθεροποιητή με πολύ μεγάλη δημιουργικότητα και φαντασία ε, αν θα βάλουμε και άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μείωση των αποθεματικών, με ε, τις ανεξόφλητες ε, φυλές. Προτείνω με το, στο Ράιμερ και το είδαμε και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα δύο κριτήρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή σύγκριση του περασμένου τριμήνου με βάση μια δεκαπενταετία και τους δείκτες της ανεργίας και μετά αν από τη μια χρονιά στην άλλη, στο ίδιο τρίμηνο, έχει αυξηθεί η ενεργεία κατά 1%. Είναι καλά τα κριτήρια αυτά για την ενεργοποίηση, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Από την άλλη, ανοίγει μια νέα συζήτηση που είναι η αποτελεσματικότητα ίδια των αυτόματων σταθεροποιητικών, χωρίς να επιστρέψουμε σε μαθήματα ε, Ιδεολογία ή πεδαγωγική ή τέτοιε συζητήσει φιλοσοφικέ τίθε το ερώτημα ε, όταν έχει αυτόματο σταθεροποιητή είσαι αποτελεστικό ε, όταν δράσει τη ζήτηση ή όταν δράσει την προσφορά όταν προσανατολίζει αυτή Η Ευρωπαϊκή τιθεται το ερωτημα οταν θέλει αποτελεσματικος οταν δρασει τη ζητηση η οταν δρασει την προσφορά με μία παρέμβαση για να στηριχθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Εμείς όμως τι διαπιστώνουμε, ότι υπάρχουν ήδη εργαλεία για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, τα οποία δεν είναι ακριβώς προσαρμοσμένα στην Ευρωζώνη ε, και υπάρχουν και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αλλά ε, από την άλλη, αν στηρίξει τη ζήτηση, ή μάλλον για τη στήριξη της ζήτησης, δεν έχουμε κανένα μηχανισμό αυτή τη στιγμή και χωρίς να αποκαλύπτω τίποτα τεράστια μυστικά που είχα σε κάποιες συνομιλίες εν ώψη της εκπόνησης της έκθεσης, θέλω να σας πω ότι συζητήσαμε με τον Όλαφ Σόλτς, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Και είπε ότι δεδομένης κατάσταση στη Γερμανία, όταν κοιτάει και μελετάει τι επέτρεψε ε, στη Γερμανία να περάσει καλύτερα την περίοδο αυτή της κρίσης από όλα τα κράτη-μέλη ήταν η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα πλεονάσματα και βεβαίως να ε, εξακολουθεί να λειτουργεί ο αυτόματος σταθεροποιητής του επιδόματος ανεργίας χωρίς να, επηρεάσει, να επηρεαστεί και μετά μπόρεσαν να φτιάξουν μηχανισμούς στήριξης ε, Nous devons euh, ouvrir cette discussion. Για τα επιδόματα ανεργίας βραχίας διάρκεια. Έχουν γίνει προτάσεις από τα διάφορα κράτη-μέλη. Και τα ξέρουμε αυτά, Ράιμερ είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένα από πανεπιστημιακά έγγραφα, βιβλιογραφία, από διεθνείς διασκέψεις και αξίζει τον κόπο να τα διερευνήσουμε. Στην πρότασή μας λοιπόν τι κάνουμε. Έχουμε και μια σειρά από στοιχεία που είναι σημαντικά για τη συζήτηση και θα τα αναφέρω εν συντομία. Τη δημιουργία ε, ενός τμήματος αυτού του μέτρου, το οποίο δεν είναι ακριβώς αντιγραφή, αλλά υπάρχει μια διευκόλυνση ε, για ε, το ισοζύγιο πληρωμών για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Δηλαδή, τι προτείνουμε. Όταν ένα κράτος μέλος μπαίνει στην Ευρωζώνη, τα χρήματα που υπάρχουν σε αυτό το αποθεματικό, σε αυτή τη διευκόλυνση ισοζυγίου πληρωμών, να μεταφέρονται για να ενισχυθεί αυτό το μέσο. Στην πρόταση όμως Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Τι γίνεται όταν το 30% των κονδυλίων του Ταμείου αυτού, το αποθεματικό, έχουν ήδη απορροφηθεί. Τι σημαίνει αυτό. Ένα κράτος μέλος ε, μπορεί να ε, ενισχυθεί ε, με ένα ποσό που έχει ανώτατο όριο τα 9 δις. Όταν έχει εξαντληθεί αυτό, τι γίνεται. Μπορεί να συνδεθεί με τον μελλοντικό μηχανισμό σταθεροποίησης. Δεν θέλω να μακρηγορήσω και να σας κουράσω. Έχω βάλει, νομίζω, τις βάσεις για τη συζήτηση και μπορούμε εκεί να αξιοποιήσουμε τη συζήτηση για να εξισορροπήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θέλει να υποστηρίξει τη δημόσια επένδυση, αλλά εμεί θέλουμε να το στρέψουμε περισσότερο στη στήριξη της ζήτησης και όχι της προσφοράς. Και ένα ε, σύστημα αντασφάλισης ουσιαστικά της ε, ανεργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές. Και τώρα πρώτος ο κύριος Σάντος Ιέιντερ εκ μέρους του. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν έσκασε η κρίση, αν είχαμε ακριβώς αυτό το μέσο σταθεροποίησης, ε, μάλλον δεν θα είχαμε τις τόσο αρνητικές επιπτώσεις ε, από αυτές που ζήσαμε. Δηλαδή, το να έχει ένα τέτοιο εργαλείο και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που θα πρέπει να αξιολογήσουμε πάρα πολύ θετικά. Με τι όποιε αδυναμίες και καθυστερήσει γιατί είμαστε δέκα χρόνια μετά. Αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και ο κύριο Μπέγκε και η κυρία Μπεραέσσα για βελτιώνουν ουσιαστικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το χρειαζόμαστε αυτό το μέσο. Βεβαίως, για τους εξή δύο λόγους. Πρώτον, προφανώς για περίοδους κρίσης, για να μπορούμε να το ενεργοποιούμε και να μπορούν να συνεχίσουν οι επενδύσεις να χρηματοδοτούνται. Αλλά το δεύτερο είναι ότι στέλνουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα στις αγορές και προς τα έξω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμαθε από τις κρίσεις και κινητοποιεί ή ε, ε, στείνει εργαλεία για να αντιμετωπίσει την επόμενη κρίση, η οποία θα έρθει. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά θα τη βρούμε μπροστά μας και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αργούμε λίγο γιατί <laughs> το καλό το πράγμα αργεί να γίνει, αλλά αντιδρούμε, εν πάση περιπτώσει. Ποιο είναι το εκ των όνων κάνευ, να είναι αυτόματος ο σταθεροποιητής. Αν δεν μπει αυτόματος χαρακτήρας, δεν θα έχει την ε, αποτελεσματικότητα που οφείλει. Και το χειρότερο ποιο είναι, 30 δις για όλη την Ευρωζώνη. Καλά, σιγά τα λεφτά. Ούτε έχει και τεράστιο αντίκτυπο. Αλλά μπορεί να αυξηθεί η πρόταση. Ένα μικρό δημοσιονομικό σχόλιο. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το, ε, το μέσο αυτό είναι εκτός ε, των οροφών του δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά θα πρέπει να εντάσσεται στην οροφή των ιδίων πόρων. Όταν ορίσουμε τις ποσότητες και τα ποσά μάλλον, δεν θα πρέπει να μειωθεί το PVP, αλλά να αυξηθούν οι διπόροι. Καλά, αυτό ήταν ένα μικρό σχόλιο προπολογισμού. Λοιπόν, το καλύτερο είναι αυτοματοποίηση, το χειρότερο είναι το ποσόν και αυτό που λείπει και συμφωνώ με τα όσα έλεγε προηγουμένως η κυρία Μπερές, είναι η ασφάλεια της ανεργίας. Για πρώτη φορά έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε ε, την ασφάλεια και αντασφάλιση της ανεργίας. Όλο και περισσότερες χώρες το βλέπουν αυτό ευνοϊκά και το Κοινοβούλιο θα διέπρεπε μέγα σφάλμα εάν δεν τα έβαζε αυτά στο συγκεκριμένο κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μουρεσάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Σε πρώτη φάση θέλω εκ μέρου τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να ευχαριστήσω του δύο συνεισηγητέ, Μπερέ Μπέγκε, για την δουλειά του που δεν έχει σταματήσει και που ξεκίνησε από πέρσι με την δημοσιονομική δυνατότητα της ε, Ευρωζώνης που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Κατά πρώτον να πω ότι εκτιμώ το γεγονός ότι οι συνάδελφοι ρητός καλούν στην έκθεση για τακτική υποβολή εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο σε σχέση με την εξέλιξη του μηχανισμού. Αυτό θα πρέπει να το επιδιώξουμε, έναν ισχυρότερο ρόλο του Κοινοβουλίου σε όλο αυτό το νέο σχήμα. Επίσης, ε, συμφωνώ με την αιρεσιμότητα. Η αιρεσιμότητα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, να είναι μικροοικονομική, να είναι μικροοικονομικά τα κριτήρια δηλαδή και με περισσότερο να δώσουμε και τις λεπτομέρειες. Υπάρχει όμως εδώ και ένα σημαντικό πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή η αιρεσιμότητα θα πρέπει να έχει να κάνει με το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και το κράτο δικαίου και να μην ε, μπορεί να βοηθηθεί μια χώρα που είναι στη δικασία του άρθρου 7. Αυτό θα πρέπει δούμε. Είναι ένα στοιχείο άκρο πολιτικό και θα πρέπει να σκεφτούμε τι επόμενε εβδομάδε αν θα το προκρίνουμε ή όχι. Ε, πέραν αυτών, ήθελα να επιμείνω σε κάποια σημεία που θα θέλαμε να το αναλύσουμε καλύτερα με τους συναδέλφους και τους εισηγητές και χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα θέμα σύγκλησης. ένα κώδικα μάλλον σύγκληση, ο οποίο καλό είναι να υπάρχει. Την καλωσορίζω την ιδέα, αλλά δεν θέλουμε να αντικαταστήσει την υπάρχουσα δημοσιονομική νομοθεσία. νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι κάτι το πρόσθετο σεβασμό του κώδικα αυτού σε σχέση με του κανόνε. Δηλαδή, μια χώρα, εάν έχει δυσκολίε, θα πρέπει να ε, εξετάζεται κατά πόσο σεβάστηκε του κανόνε, όχι αν κάποιον έχει παραβιάσει. Επίσης ο κώδικας των κανόνων θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Κριτήρια τα οποία γράφεται να υπάρχουν σε αυτόν τον κώδικα της ε, και να είναι ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει τη λογική ότι οι πληρωμές και οι επιδοτήσεις για τις υποδομές θα πρέπει να υπόκεινται στο κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα κονδύλια. Αυτή η προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των κονδυλίων έχει διαγραφεί από τους συνεισηγητές. Πώς θα ξεκινούν ε, οι πληρωμές όμως αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, αν δεν είναι διαθέσιμες. Εγώ καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι ε, προφανώς για να γίνουν πληρωμές πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο χρήμα. Ε, επίσης υπάρχει και η ιδέα του μηχανισμού ασφάλειας, ασφάλισης. Αυτό το ε, ήταν κάτι το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο όταν συζητήσαμε για την έκταση αυτή και δεν υπήρξε καμία πλειοψηφία για ένα μηχανισμό ασφάλισης. Άρα δεν μπορούσαμε τότε να εγκρίνουμε. Τι άποψη έχουν λοιπόν τώρα οι εισηγητές και γιατί διαγράψατε το στοιχείο του, της οικειοθελούς συμμετοχής σε αυτό το μηχανισμό. Αυτό το διαγράψατε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το τελευταίο στοιχείο που ήθελα να φέρω στην προσοχή σας είναι το θέμα του όγκου, της ποσότητας. Ε, έπρεπε να περιοριστούμε στα 30 δις. Ε, η... Τελικά από πού θα έρχονται αυτά τα χρήματα και μετά το ε, οι αρχέ τι οποίε θέλω να επιμείνουμε είναι η ξεκάθαρη ρεσιμότητα, οι περιορισμοί και ξεκάθαροι ορισμοί σε ό,τι αφορά τον κώδικα συγκλήση και την συμμόρφωση με του υπαρχόντες δημοσιονομικού κανόνες. Ευχαριστώ. Ε, η συμμόρφωση υπάρχει. Το βλέπετε. Δεν είναι κάτι που λείπει. Λοιπόν, Bernd Δεν το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό θέλω να μιλήσω στα γερμανικά. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Και το μέσο αυτό μπορεί να είναι τεχνικά θαυμάσιο, αλλά έχει λανθασμένη αφετηρία. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς είναι πάρα πολύ απλά το νόμισμα που λέγεται ευρώ, το οποίο έχει λάθος σύνθεση και γι' αυτό θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί πολλά πράγματα. Βεβαίως κάνουμε άλλα τα οποία δεν λειτουργούν και συνεχώς εφευρίσκουμε νέα μέσα. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι να αναφερθούμε στο πρόβλημα το ίδιο που λέγεται ευρώ για να γλιτώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Και δίνω τον λόγο στον συνάδελφο τον Μπέρντ Λούκε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκε. Ο συνάδελφος ε, μου άφησε άλλο ένα λεπτό γιατί υπάρχουν πολλά που πρέπει να πούμε. Η νομοθετική αυτή πρόταση ε, αποκλίνω λίγο από την διπλωματική γλώσσα των συναδέλφων, είναι η χειρότερη που έχω διαβάσει ποτέ από την Κομισιόν. Δεν την έχει σκεφτεί σωστά. Ε, πλησιάζει σοσιαλιστική κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία και είναι τελείως απλά ψευδής και ε, δεν το διόρθωσαν οι δύο συνάδελφοι. Κύριε Μπέγκε, πραγματικά σας εκτιμώ προσωπικά, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει πουθενά η υπογραφή του ΕΛΚ. Αναγνωρίζω όμως ε, την υπογραφή των ε, σοσιαλδημοκρατών. Να σας πω γιατί είπα ότι είναι μια έκθεση ψευδής. Μας λέει ότι έχουμε ένα μηχανισμό επενδύσεων για μεγάλους ασύμμετρους κρατασμούς. Αλλά η αιτιολόγηση είναι η οικονομική κρίση, η οποία ήταν ξεκαθαρά συμμετρικός κραδασμός. Επηρέασε αρνητικά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρξε κάποια ασυμμετρία. Το ότι εδώ πέρα μιλάμε για ασύμετρο σοκ και στα εκτιμώντας μάλιστα αναφέρεται ρητός η οικονομική κρίση είναι ψευδές γιατί ε, ακριβώς έχουμε την πολιτική συνοχής ε, και Εκεί έχουμε χρησιμοποιήσει αυτήν την αιτιολόγηση. Αλλά η οικονομική κρίση δεν ήταν κάτι τέτοιο, δεν ήταν ασύμετρος κραδασμός. Καλό είναι λοιπόν να ορίσουμε κάπου και να, δούμε τον ορισμό του ασύμετρου σοκ. Επίσης, είναι κατά της οικονομίας της αγοράς γιατί δεν θα υπάρχει ένας μηχανισμός των επιτοκίων, αντιθέτως θα υπάρχει επιδότηση των επιτοκίων. Μιλάμε για κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία γιατί μιλάμε για αυτοματισμό και δεν υπάρχει καν η πρόθεση να μιλήσουμε για την αποδοτικότητα των επενδύσεων. Αρκεί μόνο να δώσουμε λεφτά χωρίς να δούμε εάν θα είναι κερδοφόρες αυτές οι επενδύσεις. Αυτό δεν έχει ούτε μία σχέση με η οικονομία της αγοράς. Επίσης δεν συμφωνώ με τον κύριο Μπέγκε όταν είπε και, είπε και η κυρία Μπερέ κάτι ανάλογο ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας μηχανισμός ενεργοποίησης τον οποίο έχουμε σκεφτεί προσεκτικά. Αντιθέτως, αν δούμε την ε, ανεργία τότε το θέμα μας δεν είναι αντίδραση στο σοκ, αλλά η δυνατότητα αντίδρασης μιας οικονομίας. Και αν είναι ευέλικτη περισσότερο ή λιγότερο, σημαίνει ότι μια αγορά, μια ε, χώρα, μια οικονομία με πιο ευέλικτη αγορά εργασίας θα αντιμετωπίσει καλύτερα την κρίση σε σχέση με μια χώρα η οποία είναι πιο ε, άκαμπτη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ο μηχανισμό αυτό θα απευθύνεται σε αυτέ τι χώρε οι οποίε δεν έχουν κάνει τι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει που θα έπρεπε. Δηλαδή, εδώ πέρα δημιουργούμε λάθο κίνητρα. Και τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, προφανώς δεν έχουμε σκεφτεί ποια είναι η σχέση μεταξύ τη προωθηση δημοσίων επενδύσεων που υποτίθεται επίση θα έπρεπε να έχουν μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία που επίση δεν έχει καθοριστεί και των ε, επενδύσεων των ιδιωτικών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και εδώ πέρα θα δημιουργήσουμε ένα φαινόμενο crowding out. Θα διώξουμε δηλαδή ε, επενδύσεις. Έχουμε λοιπόν ένα μέσο που είναι κατά της ε, ελεύθερης αγοράς και είναι ψευδές. Γι' αυτό τα είπα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι σοσιαλιστικό, γιατί ε, με τη λογική σας το Δέλτα είναι σοσιαλιστικό, η ΕΠΑ είναι σοσιαλιστική χώρα και όλες οι χώρες που έχουν αυτόματο σταθεροποιηθεί είναι σοσιαλιστικές. Ζούμε σε κόσμο σοσιαλιστικό λοιπόν, χωρίς να το ξέρουμε. Μα κάτι μάθαμε και σήμερα. Λοιπόν, Ούρμα Σπάιτ από την Άλντε, από ο Τρεμόσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ. Και σε σχέση με αυτά που είπα προηγουμένως στην προηγούμενη συζήτηση, εμείς κάνουμε μια συζήτηση ε, λογική ε, στους φιλελευθέρους. Όπως ξέρετε, έχουμε διάφορες τάσεις ε, από διάφορες χώρες προερχόμενοι και διαφορετικούς πολιτισμούς. Έχουμε και διαφορετικές απόψεις για κάποια θέματα. Ε, ο συνάδελφος Μούρες, αν το είπε προηγουμένως, θα πρέπει να συζητήσουμε και τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Υπό ποια ανένεια. Η έκθεση αυτή What are we here in terms of... Ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και κάποιο καταμερισμό κινδύνου και περιορισμό κινδύνου, μείωση. Αυτό είναι το πλαίσιο το γενικότερο. Πολλά μέλη της ομάδας μου καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στις διαφορετικές μεταφορ... μεταρρυθμίσεις συγγνώμη, και τη συμμόρφωση στο σύμφωνο σταθερότητα. σταθερότητας. Να σας εξηγήσω κάτι. Μπορεί να θυμάστε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγα χρόνια ο πρόεδρος ομάδα, δι, ε, Ομπάμα διέσωσε τη General Motors που είναι αυτοκινητοβιομηχανία. City of Detroit. Αλλά δεν διέσωσε ο πρόεδρος Ομπάμα την πόλη του Detroit. Γιατί στο τέλος του 19 στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ε, σφυριλατούσαν την ένωση τους ε, έλεγαν θα έχουμε ένα μοσπονδιακό ε, ε, χρέος. Ε, συμφώνησαν λοιπόν όταν στείναν αυτό το σύστημα ότι δεν πρόκειται να ε, σώνουν με δημόσια χρήματα ε, πόλεις και πολιτείες. Άρα όταν υπάρχει αυτό το θέμα της αιρεσιμότητας, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Δύο λεπτά και δεν τα ξεπερνάω, όπως και την περασμένη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, for the Greens, Ο Γιώργη Σολέ από τους Πρεσίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την αδειά σα ε, θα πάρω και τα δύο λεπτά του συναδέλφου του κυρίου Λαμπέρτ. Είναι επιχορήγηση, δάνειο, τι είναι. Επιδότηση. Ε, είναι μια χάρη, χάρη από τον συνάδελφο. Ε, στην υπηρεσία του λαού. Mm. Ήδη 20 δευτερόλεπτα πέρασαν όμως. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε πέντε σημεία το πρώτο φορά το μέγεθο και εμεί θεωρούμε ότι 30 δισεκατομμύρια για την περίοδο 21-27 είναι λίγα και δεν επαρκούν. Αν ο στόχος είναι να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέσο να αντιμετωπίσει τους ασύμετρου κραδασμού. άρα προτείνουμε το επίπεδο να είναι τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ τη Ευρωζώνη. 120 δισεκατομμύρια δηλαδή. Που σημαίνει ε, πάλι το διπλάσιο από αυτό που προτείνουν οι συνεισήγητες στην τροπολογία 19. Επιπλέον, είμαστε υπέρ ε, του να προσθεθούν ε, ή να δοθούν επιχορηγήσεις αντί για δάνεια, καθώς θα έχουν περισσότερο σταθεροποιητικό χαρακτήρα. Δεύτερον, για την αιρεσιμότητα, πέρα από τη συμμόρφωση με του ουσιονομικού κανόνε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπουν κάποιοι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί όροι για την επιλεξιμότητα, παραδείγματο χάρη η επίτευξη των στόχων του 2020. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου. Τρίτον για τους δείκτες θεωρούμε ότι οι δείκτες ε, που θα χρησιμοποιηθούν ως ε, κριτήριο θα πρέπει ακριβώς να τους επεξεργαστούμε. Το να έχουμε δύο σορευτικές ε, συνθήκες είναι πολύ περιοριστικές, ειδικά για τις χώρες που είχαν τα τελευταία 16 τρίμηνα τεράστια ανεργία. Για μας ένας όρος αρκεί για να υπάρχει πρόσβαση στο μέσο. Ε, θα πρέπει να αποκλείσουμε αλλιώς ε, κράτη-μέλη ε, τα κράτη-μέλη με ανεργία πάνω από το όρο της Ένωσης δεν θα πρέπει να πληρούν τους δύο όρους. Κατόπιν, για την φύση των επενδύσεων, βεβαίως η ομάδα μας θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρασίνισμα και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπουν και κάποια κριτήρια κοινωνικά και απασχόλησης. Και τέλος, για το δημόσιο χρέος θεωρούμε ότι τα ποσά που παρέχει το μέσο αυτό στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξαιρούνται από τους υπολογισμούς δημοσίου χρέους. με το σκεπτικό ότι θα πάνε σε επενδύσεις για δημοσίες υποδομές ε, και αποτελούν ε, πρωτογενή σχηματισμό κεφαλαίου. Σας ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ υπάρχουν ομιλητές. Ε? Όχι. Η FDD δεν βλέπω. Η ΕΝΕΦ. Ο κ. Τζάνι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ συνοπτικά. θα Πρέπει να ε, δούμε τα σημεία της πρότασης αυτής, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι πρόταση που θα λύσει προβλήματα στην Ευρωζώνη. Μου φαίνεται ότι είναι μια από τις πολλωστές, πολλαπλές απόπειρες που έχουν γίνει στο παρελθόν να λύσουμε ένα πρόβλημα διαρθρωτικό. Να αντιμετωπίσουμε με μια σπιρίνη όγκο, ε, καρκίνο. Τρία στοιχεία σημαντικά. Αυτό που είπε και ο συνάδελφος Λούκε, ότι ένα εργαλείο αυτής, αυτού, αυτής της φύσης δεν μπορεί να απορροφήσει τα συμμετρικά σοκ. Όμως δεν μπορεί να απορροφήσει και δεν μπόρεσαν και τα ανάλογα να απορροφήσουν ε, το σοκ της μεγάλης κρίσης, που δεν ήταν ε, συμμετρικό. Ήταν ε, κάτι που έπληξε ολόκληρη την Ήπειρο. Και έπειτα, για άλλη μια φορά, με ένα εργαλείο ε, χρηματοδοτικού χαρακτήρα προσπαθούμε να λύσουμε μέρος του προβλήματος πρόβλημα που σε μια χώρα κανονικών συνθήκων έπρεπε να επιλύεται με νοσματικές πολιτικές. Οι κεντρικές τράπεζες ε, στην εντολή τους ε, έχουν το καθήκον να παρακολουθούν το επίπεδο της απασχόλησης και να αντιδρούν όταν αυτό δεν είναι στο ύψος των προσδοκιών. Εμείς εδώ προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με ένα ακόμα εργαλείο που είναι αναποτελεσματικό Επίσης, η αιρεσιμότητα. Το να συνδυάσουμε, να προβλέψουμε τέτοια αιρεσιμότητα για αυτό το εργαλείο θα το κάνει αναποτελεσματικό για άλλη μια φορά. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη θα διστάσουν, θα επιφυλαχθούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό. Ε, και επίση προσπαθούμε να αυξήσουμε τι συνεισφορέ των μελών, ιδίω αυτών που τα τελευταία χρόνια ε, προσπάθησαν να στηρίξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και του ζητάμε περισσότερο χρήμα για ένα εργαλείο που ε, αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα διαφορετικά, τα δομικά προβλήματα τη Ευρωζώνη σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στο Catch the Eye. Ο κύριος Καλουέ Αμπών και ο κύριος Χιον Χώνας Ποιος άλλος? Με Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ιδέες θέλω να αναφέρω για να μην καταχραστώ του χρόνου σας. Το πρώτο που με ενέπνευσε το... η ε, τοποθέτηση του κυρίου Λούκε για την Ευρώπη ολόκληρη και την Ευρωζώνη ήταν συμμετρικός κραδασμός η κρίση, αλλά εντός της Ευρωζώνης ήταν ασύμετρες οι συνέπειες και εκεί θα πρέπει εμείς να παρέμβουμε. Έλεγε ο συμπατριώτης μου, ο Ισπανός από την Άλντε, ε, ε, μίλησε για το Τιτρόιτ, αλλά ε, και η Καλιφόρνια όταν είχε καταχρεοκοπήσει ε, δέχτηκε βοήθεια. Ήρθε ένας ομοσπονδιακός ε, ελεγκτής και έγινε παρέμβαση μέχρι και για να αγοράζει μολύβια ο κυβερνήτης στην Καλιφόρνια. Και τελειώνω. Υπάρχει και η, ε, άποψη της απασχόλησης. Ακόμα και για δεοντολογικούς λόγους πρέπει να καταγγείλουμε το γελίο ποσό. Ξέρω ότι είναι γελίος ο προπολογισμό για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό έχουμε και γελίους προϋπολογισμούς επιμέρους. Αλλά να θεωρήσουμε ότι τα μισά όσα δόθηκαν στην Ιρλανδία στην τελευταία κρίση θα αποτελέσουν αυτόματο σταθεροποιητή για την επόμενη, ε, είναι γελίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να το καταγγέλουμε μπορούμε. Ξέρω ότι έχετε ζητήσει να είναι αυτόματη η ενεργοποίηση. Εμένα με ανησυχούν και οι ε, κοινωνικές συνέπειες ε, στην ε, ζήτηση μπορούμε να παρεμβούμε ως εξής, να βελτιώσουμε ή να διευρύνουμε τους κοινωνικούς παράγοντες, δείκτες. Ας πούμε, όταν επιδεινώνεται συνεχώς η φτώχεια. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συζητητές. δικτες ας πάρα πολλά από τη δουλειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χώνας, σε ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι το σημαντικότερο στην πρόταση αυτή είναι ότι ο σταθεροποιητής ε, θα πρέπει να είναι πραγματικά αυτόματος, όπως είπε και η Περβάνς Μπερές. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, όταν το βάζει σε σύστημα ε, εγγύησης ε, των επενδύσεων, οι επενδύσεις τους από τη φύση τους έχουν περίοδο ρήμανσης πολύ μακρύτερο. Ετοιμάζεται ένα σχέδιο, μελετάτε, υλοποιείτε και τελικά έρχεται η επένδυση χαιρετίσματα ε, για τον αυτόματο χαρακτήρα αν το προσανατολίσουμε στις επενδύσεις. Διότι προφανώς οποιαδήποτε σύστημα εγγύησης επενδύσεων θα έχει μια χρόνο καθυστέρηση από τη στιγμή που ενεργοποιείται μέχρι τη στιγμή που επενδύεται ε, το χρήμα αυτό. Το είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένω, οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτες, ότι για να εγγυηθούμε αυτό τον αυτόματο χαρακτήρα, καλό θα ήταν να μην χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις, αλλά την κατανάλωση, που αυτό κάνει αυτόματο το σύστημα. Και αυτό θέλουμε εμείς να μεταρρυθμίσουμε ε, το σύστημα σε ένα σύστημα προστασίας της ανεργίας Εξού και η αυτοματοποίηση του συστηματο. Αν από την άλλη θέλουμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα σταθεροποιεί βάσει των επενδύσεων, ε, τότε θα έπρεπε να διατηρήσουμε στο πρόγραμμα EU Invest ή e Invest EU κάποια αντικυκλικά προφίλ χρησιμοποιώντας την εγγύηση ε, τους πολλαπλασιαστές έτσι ώστε το EU Invest να ασχολείται με τις επενδύσεις που κατά τα άλλα είναι ιδιωτικές επενδύσεις για να κινητοποιούνται πιο γρήγορα και από την άλλη αυτόματο σταθεροποιητής να προορίζεται στην κατανάλωση και μόνο για να έχουμε αυτή την αντικυκλική ε, συνέπεια και λειτουργία που φιλοδοξούμε. Ευχαριστώ, Ζαν Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές μας που εδώ και τρία χρόνια με ιδιαίτερη ε, αποφασιστικότητα επιδιώκουν να ετοιμάσουν μια τέτοια, αυτή την πρόταση. Είναι άοκνες προσπάθειές τους και η επιμονή τους με εκπλήσει, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της δεν μας ικανοποίησε πλήρω. Για άλλη μια φορά ε, προτείνεται ένα εργαλείο που δεν είναι στο ύψος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, το κοινό νόμισμα, η κοινή νομισματική πολιτική δεν συνδυάζεται με τις πολλαπλές εθνικές πολιτικές. Αυτό που εδώ συζητούμε είναι η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης η οποία παραμένει πολύ εύθραυστη με σοβαρούς κινδύνους και τα 30 δις δεν είναι στο ύψος των ε, κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε αύριο. 30 δις είναι πίνατς, είναι σαχλαμάρες, τίποτα. Ε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι με τις πολιτικές μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Συγχαίρω λοιπόν τους δύο συνεισηγητές, έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά εδώ απευθύνουμε έκκληση στους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων για να αλλάξουν λίγο το software που χρησιμοποιούν. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι μας έχουν μείνει μόλις πέντε λεπτά, οπότε δεν θα μιλήσω γιατί με κάλυψε ο συνάδελφος. Όσον αφορά λοιπόν την αποτελεσματικότητα, την τεχνική πτυχή της δυνατότητας να απορροφηθούν ασύμμετροι κραδασμοί, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ε, το επίδομα ανεργίας ε, είναι ο πραγματικός αυτόματος ε, σταθεροποιητής. Και μετά μπορούμε βεβαίως να μιλήσουμε για σήμανση κτλ. Αλλά δεν είναι καθόλου ασύμβατο αυτό αλλά θα ήθελα οι συνεισηγητές να σκεφτούν ε, ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να δούμε τον στόχο που φαίνεται να έχουμε κοινό. Κομισιόν, σύντομα όμως, γιατί μετά θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους δύο συνεισηγητές για την διαφωτισμένη τους ε, προσέγγιση προς την πρωτοβουλία αυτή της Κομισιόν έχουν αντιληφθεί το τι διακυβεύεται. Αυτό είναι το πρώτο συγκεκριμένο βήμα των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για έναν μηχανισμό συλλογική αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν ασύμετρους κραδασμούς ε, καθώς έχουν, ε, δεν έχουν πλέον την δυνατότητα που τους παρήχε η συναλλαγματική ισοτιμία. Πρόκειται δηλαδή για κάτι το οποίο θα βοηθήσει χώρε οι οποίε έχουν χρηστή διαχείριση όταν αντιμετωπίζουν κάτι εκτό του ελέγχου του πριν βρεθούν σε ανάγκη να χρειαστούν ένα δομημένο πρόγραμμα βοήθεια. Αυτό είναι ο στόχο. Θα συμβούν αυτοί οι κρατασμοί, έχουν ξανασυμβεί, καταραίουν ε, συχνά και οι τιμέ των ακινήτων. Ε, έχουμε ε, άλλε χώρε στην Ανατολική Ευρώπη που βρίσκονται σε μια δύσκολη γειτονιά Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε και το σχέδιο έκθεσης ορίζει, θα λέγαμε, το πλαίσιο και για αυτό το οποίο είπατε για το επίδομα της ανεργίας νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον ε, διαδίδεται στις πρωτεύουσες ε, και υπάρχουν κάποιες πρώτες ε, κρούσεις στο Συμβουλίο Κομισιόν. Οπωσδήποτε θα το δει το θέμα επικοδομητικά. Θα προσπαθήσουμε να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση Πρέπει να σεβαστούμε την νομική βάση, να αποφύγουμε τον να εστιάσει το θέμα στα επιδόματα ανεργίας ε, και να μην επηρεάσει έτσι τον αυτοματισμό και την γρήγορη χρήση και να μην μπουν όροι ε, στα εθνικά συστήματα επιδόματος ανεργίας. Αλλά υπ' αυτούς τους όρους θα ακολουθήσουμε το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη στην κατεύθυνση που αυτά θέλουν. Ε, σύντομα για το μέγεθος του προϋπολογισμού. Δεν είναι αυτό το μόνο μέσο που έχουμε για την αντιμετώπιση της κρίσης αφορά τη σταθεροποίηση των δημοσίων επενδύσεων πριν ε, πληγεί μια χώρα από την κρίση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στο ΠΔΠ, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούσε να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στην σταθεροποίηση μέχρι και ενός 10% των δημοσίων επενδύσεων. Είναι μέρος της λύσης και είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση που πρέπει να πάμε. Και τέλος, Καλωσορίζουμε τις ε, δηλώσεις ε, της κυρίας Μπερές για τους όρους ενεργοποίησης, ε, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει ο μηχανισμός αυτός να είναι στόχευμένος σε αυτούς οι οποίοι το αξίζουν στις χώρες με την καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση, οπότε θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του να προωθήσει αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, ο κύριος Μπέγκε. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ο κύριος ε, Λούκε έχει ε, δίκιο, δεν ήταν ενωμένη ομάδα του ΕΛΚ, αλλά κατά πλειοψηφία ήταν ε, στο πλευρό μου και χάρηκα γιατί αυτό ήταν το σωστό. Κοιτάξτε, όταν μιλάτε για ψεύδι, εγώ ευθυγραμμίζομαι με το ΔΕΛΤΑ με τον Κλάους Ρέγκλινγκ που είναι αναμφισβήτητα ειδικό και με τον καθηγητή Φιούστ του Ινστιτούτου του Μονάχου, με τον κύριο Ντιμάουρο, δηλαδή με ε, ειδικού εγνωσμένου ε, κύρους. Δεν είμαι τόσο ειδικό στα οικονομικά, αλλά θυμάμαι ότι τα οικονομικά δεν είναι θετική επιστήμη, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. του Μορεσάν, δείτε τους ορισμούς. Λέει ότι υιοθετείται με βάση την τακτική νομοθετική διαδικασία. Πρέπει να μπει, ναι, το διατυπώσαμε έτσι, υπάρχει μια σχέση και νομίζω ευχαριστώ να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς ε, ορίσαμε ως ενεργοποιητή το επίπεδο της ανεργίας, ε, το, γιατί το Συμβούλιο είπε ότι εάν θέλουμε να έχουμε έναν αυτόματο ενεργοποιητή, αυτός είναι ο καλύτερος και ο σαφέστερος. Αλλιώς μπορούμε να διατυπώσουμε 10 ε, πτυχές ε, και δεν θα λειτουργεί τίποτα. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσω και πάλι, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς ε, εδώ πέρα, με τις τροπολογίες, δεν είναι, δεν σημαίνει ότι δίνουμε εξοδότηση λευκό για μια ασφάλιση ανεργίας. Διακόπτεται η διερμηνία, ρωτάει ο κύριος Μπέγκε. Ε, πρέπει να σταματήσει η διερμηνία εδώ, τελειώνει η διερμηνία με βάση το πρόγραμμα. Οι διερμηνείς έχουν και άλλη συνεδρία στη συνέχεια. Which was presented also from uh, Minister Scholz. Um, yes, you may discuss it, but it was something we, at this point, didn't want to have as amendments to go in what direction, because there we have different differences